την αρμόδια νομική επιτροπή ε, από ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ε, την Ελευθερία και Δημοκρατία έχουν υποβληθεί αιτήματα για ορισμούς σε επιτροπές και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή εστάσεις θεωρούνται αυτοί οι διορισμοί εγκεκριμένοι. Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε